σε ιδιωτικές και κρατικές αρχές να επενδύσουν βιώσιμα με συγκεκριμένους κανόνες και κίνητρα. Συμφωνήσαμε πολύ πρόσφατα στην ταξινομία για να καθορίσουμε και να ορίσουμε επακριβώς ποιες είναι οι ε, ε, οικολογικές επενδύσεις, ποιες είναι οι βιώσιμες επενδύσεις, αυτό και για τον κρατικό και για τον ιδιωτικό τομέα. Ε, Αργότερα θα υποβάλουμε και πρόγραμμα, επανανεωμένο πρόγραμμα επενδύσεων. Επίσης, ε, θα αναθεώσουμε τους κανόνες μας σε ό,τι αφορά τις κρατικές προμήθειες. Τρίτον, δεν μιλάμε μόνο για χρηματοδότηση, έχουμε και, το, και τα συγκεκριμένα σχέδια. Οι εθνικές διοικήσεις ε, θα λάβουν τη βοήθεια εμπειρογνωμών, εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουμε, ε, <clears throat> μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για παράδειγμα, για να πετύχουν τους στόχους τους. Περνώ στο δεύτερο κομμάτι της συζήτησης που είναι ο δικός χάρτης για μια κοινωνική Ευρώπη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ε, ως για την οικονομία που δουλεύει προς συμφέρον του, ε, ε, των πολιτών θα πρέπει ε, να, να είμαστε δίκαιοι και να συμπεριλαμβάνουμε όλους την ανάπτυξή μας. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων και είμαστε δεσμεμένοι σε αυτό και το σημερινό μας ανακοίνωθεν, η σημερινή μας ανακοίνωση θέλει να μεταφράσει αυτό τον πυλώνα σε πραγματικότητα με συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό επίπεδο ε, ή και από τον ιδιωτικό ε, τομέα. Θέλουμε να μας πούν όλοι οι εταίροι ποιε είναι οι προσπάθειε που πρέπει να μπορούν να κάνουν. Θα ξεκινήσουμε μια διαβούλευση λοιπόν με του κοινωνικού εταίρου, για παράδειγμα για το ε, ε, ελάχιστο ε, μισθό, για το ελάχιστο ημερομίσθιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρόκειται να καθορίσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κατώτατο ημερομίσθιο, ούτε θα υποχρεώσουμε κάποιον να καθορίσει τέτοιο μισθό, θα σεβαστούμε τις συλλογικές συμβάσεις. Η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα απαιτεί να αλλάξουμε νοοτροπία. Ήδη κάναμε ένα πρώτο βήμα σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα λοιπόν εκ μέρου ε, του ΕΛΚ ο κύριος Σικφρίτ Μουρεσάν. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, κύριε Αντιπρόεδρε Λομπρόφσκι. σα καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστούμε που μα παρουσιάσατε τι πρωτοβουλίε Εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να χαιρετήσω τι προτάσει που παρουσιάσατε σήμερα και πιστεύω ότι αυτό ο δίκαιο μηχανισμό, αλλά και όλα αυτά που παρουσιάσατε σήμερα είναι απολύτω απαραίτητα για την επιτυχία δύο πολύ σημαντικών προγραμμάτων για το Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω να συμφωνήσουμε το των δυνατόν κατά τους πρώτους μήνες αυτού του έτους σχετικά με τον δίκαιο μηχανισμό γιατί έτσι λοιπόν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει για το πουδουπού και επίση θα καταστεί δυνατόν να στεφθεί από επιτυχία η Πράσινη Συμφωνία. Το Δεκέμβρη είδαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η Πράσινη Συμφωνία, πρέπει να πετύχει, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διευκρινίσουμε ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν τον μηχανισμό δίκαιη ε, μετάβαση. Πώ λειτουργεί αυτό και πώ πρέπει να είναι. Πρώτον, πρέπει να είναι σταθερό, να είναι πρικοδοτημένο σωστά για να ε, υπάρξει διαφορά, κυρίως ε, στις φυγήσει περιοχές. Δεύτερον, ούτε η συνοχή, ούτε η γεωργία, ούτε η καινοτομία δεν αφορούν αυτό το ταμείο. Θα πρέπει να χρηματοδοτείται με κάτι παραπάνω. Και τέλο, να έχει μακροχρόνιε προεκτάσει αποφάσεις. Αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομική ανάπτυξη, να στηρίξουμε τις επιχειρηματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην ε, επαναλάβουμε ε, τα λάθη, κυρίως αυτά που αφορούν ανθρώπους που δεν είχαν τις απαραίτητες δεξιότητες. Και τέλος, όσον αφορά τις προϋποθέσεις, πρέπει να εκταμιεύσουμε χρήματα στις χώρες, στις περιοχές, σε προϋποθέσεις που είναι αποδεκτές, να μάθουμε από την εμπειρία του InvestEU από το παρελθόν και από άλλα προγράμματα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Και τώρα λοιπόν εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Γκαρσία Πέρε, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Το περασμένο Δεκέμβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της για τη νέα πράσινη συμφωνία. Είναι φιλόδοξη η πρόταση και ακριβώς ε, στόχο έχει την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι είναι κολοσιαίο αυτό το έργο που χρειάζεται μια πραγματική μετάβαση και μετασχηματισμό των κοινωνικο-οικονομικών μας συστημάτων αλλά και του τρόπου ζωή μα. Η αξιοπιστία αλλά και η επιτυχία τη πράσινη συμφωνία, θα εξαρτηθούν από τα σχέδια χρηματοδότηση. Να δούμε όμω πώ θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον αντίκτυπο αυτού του μετασχηματισμού στι περιφέρειές μα που έχουν ενεργειακά βιομηχανικά μοντέλα τα οποία απαιτούν πιο ακριβό μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό. Τα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα πρώτα βήματα. Θέλετε να βρεθεί ένα δισεκατομμύριο, ε, μάλλον ένα τρισεκατομμύριο την επόμενη δεκαετία για να είμαστε οι πρώτοι μέχρι το 2050. Άρα ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια θεωρεί ότι το 1-3 στο οποίο φιλοδοξεί είναι ε, το ελάχιστο κλάσμα του απαιτούμενου ποσού για την ε, μετάβαση αυτή. Οι υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε ε, συστηματικά και μεθοδικά. Χρειάζεται οπωσδήποτε συζήτηση για να δούμε πού θα βρούμε νέα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη κοινωνική, οικολογική και οικονομική μετάβαση. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες έχουμε πολύ στεναρή στάση σχετικά. Θέλουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να αφιερώνει τουλάχιστον το 30% στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον όμως θα πρέπει να συζητήσουμε και για τους ιδίους πόρους που να συμπεριλαμβάνει ένα τέλος ε, από τα πλαστικά ε, να συμμετέχει η ψηφιακή οικονομία, να υπάρχει φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μια ενιαία κοινή ε, βάση ε, για τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η διπόρη. Επίσης, εμείς διεκδικούμε τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο χειρισμών στους εθνικούς προϋπολογισμούς για να ενθαρρύνουν βιώσιμες επενδύσεις. Και να γίνει αυτό το τελευταίο πραγματικότητα, προτείνουμε να μεταρρυθμιστούν οι κανόνες, οι δημοσιονομικοί, έτσι ώστε οι βιώσιμες επενδύσεις να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ελλείμματος και του χρέους ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η δίκαιη μετάβαση. Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει στην άκρη. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι σλόγγαν απλώς ε, σύνθημα. Θα πρέπει το Ταμείο Δίκαιης ε, Μετάβασης να έχει επιπλέον οικονομικούς πόρους για να μην μειωθεί η πολιτική συνοχή ούτε η κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό σημαίνει να αποκτήσουν δεξιότητες οι εργαζόμενοι έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την οικολογική και ψηφιακή μετάβαση. Επίσης θα πρέπει να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για να ε, σπάσει, να κλείσει μάλλον η ψαλίδα η ε, μισολογική και να καταπολεμήσουμε ε, την παιδική φτώχεια. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε από κοινού, με συνεργασία, αλλά και με οικονομική δέσμευση. Ευχαριστώ. Από την ομάδα Renew Europe το λόγο τώρα έχει ο κύριος Πισλάρου. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Um, <clears throat> thank you, um, Madam Chair. I uh, prea mult... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ συχνά η Ευρώπη έχει δεχθεί, ε, δεχτεί κατηγορίες γιατί δεν κάνει τα λόγια πράξη. Άλλε φορέ κατηγορείται για, να, για το ότι δεν έχει επαρκές όραμα. Σήμερα ε, βάζουμε δίπλα-δίπλα πολλά εργαλεία τα οποία εξυπηρετούν το ίδιο όραμα της ε, Πράσινης Συμφωνίας και εστιάζονται στον πολίτη. Το μήνυμα που θέλουμε εμείς να στείλουμε είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να συγκρατήσουν πως η Ευρώπη θέλει να μετατρέψει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής σε ευκαιρία. Με περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι πολίτες ε, των πιο ευάλωτων περιοχών, όπως στη Ρουμανία, των πιο φτωχών περιοχών επίσης, θα μπορούν να επωφεληθούν από πρόσθετα εργαλεία, πρόσθετη βοήθεια μέσω του Ταμείου ε, δίκαιης μετάβασης. Αυτό θα τους δώσει καινούριες ευκαιρίες και θα προετοιμάσει επίσης τους νέους ε, έτσι ώστε να αποκτήσουν έγκαιρα τα κατάλληλα προσόντα και τις κατάλληλες δεξιότητες. Επίσης θα ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διευκολύνουν αυτή την επαγγελματική κατάρτιση των νέων ιδιαίτερα σε θέματα τεχνολογίας. Πρέπει να είναι δίκαιη μετάβαση γιατί μόνο έτσι θα θα αγγίξουμε όλους τους πολίτες και θα έχουμε μόνιμα ωφέλη για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα μέσα τα οποία θα αποφασίσει η Κομισιόν και θα πρέπει σιγά σιγά να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. ο λόγος του κύριο Νίνας. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την πρόταση για ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης. Ε, κατανοώ βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση ε, Πρέπει να υπάρχει επίσης ένα απόλυτο σαφές ε, για το να μην υπάρξουν αποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων. Αυτή η πρόταση είναι ένα καλό σημείο κίνηση ε, για να βοηθηθούν κυρίως ορισμένες περιοχές έτσι ώστε να έχουν μια δίκαιη μετάβαση. Αυτό όμως που δεν υπάρχει στην πρότασή σας είναι μια σαφή ε, δέσμευση για, τις κλιματικές, για την κλιματική αλλαγή. Οι άνθρωποι χρειάζονται μια σαφή δέσμευση από κάθε μεμονωμένη περιοχή για προγράμματα απομάκρυνσης από τον άνθρακα. Ε, δεσμευτική λοιπόν αυτή η προϋπόθεση για να λάβει κανείς την ε, χρηματοδότηση από το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Γιατί αν δεν υπάρχει απομάκρυνση από τον άνθρακα, αυτό δεν έχουν νόημα και βεβαίω ε, και πρέπει να μιλάμε για χρήματα 7,5 σε 7 χρόνια σε πολλές περιοχές, άρα δηλαδή 10 εκατομμύρια αναπεριοχή ανά έτος. Αρκεί αυτό για να είναι δίκαιη μετάβαση για και κατόπιν μπορεί κανείς και να προσθέσει και τη χρηματοδότηση από άλλα ταμεία. Αυτό όμως είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν θέλουμε να μετακινηθούν κονδύλια από μία περιοχή σε άλλη περιοχή. Και αν τα πολλαπλασιάσει κανείς με ιδιωτικέ επενδύσεις, αλλά κύριε Τίμερμαν, σε γνωρίζουμε ότι ε, δεν είναι τα 100 δις, αλλά είναι κατ' ουσίαν 7,5 δις κατ' ουσίαν ε, προσπαθούμε να προβάλλουμε το θέμα με τρίκο όμως ε, και εγώ δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμφανίζεται ως ο μάγος που βγάζει από το καπέλο του να έχουμε ένα καλύτερο ταμείο με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε οι ανθρακορίχοι να μην είναι στο έλεος ε, κάθε 7 χρόνια των διαπραγματεύσεων για το πουδουπού. Εμείς θα τα στηρίξουμε αυτά αν πραγματικά υπάρχει μια σαφής και δίκαιη μετάβαση με συγκεκριμένο πρόγραμμα απομάκρυνσης από τον άνθρακα για όλες τις περιοχές όπου σήμερα υπάρχει άνθρακας. Πολύ ωραία. Τώρα ε, ο κύριος ε, Αντώνιο Νταρέ ε, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Χίλια δις για τα επόμενα χρόνια αυτό είναι το πρόγραμμα έτσι ώστε να επιτευχθεί η κλιματική οδετερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050. Γνωρίζουμε τον προπλησμό χίλια δις. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι από πού θα έρθουν όλοι αυτοί οι πόροι ε, και ίσως ε, να πρέπει να περιοριστούν τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να λύσουμε και άλλους δύο ε, γόρδιους δεσμούς, ε, το πώς θα μπορέσουμε να διανύμουμε αυτούς τους πόρους για να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση από τα κράτη. Μιλάμε για ένα ταμείο, για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να είναι μόνο ένα σύνθημα, αλλά συγκεκριμένες πράξεις που θα φαλίσουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για τις οποίες δεν γίνεται καθόλου λόγους σε αυτό το πρόγραμμα των επενδύσεων. Ευχαριστώ από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώχαν Πανόβερφελτ. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροποι, μόλις επιβεβαιώσατε αυτό που είχα φοβηθεί το Δεκέμβριο πολύ θελησιοκρατικό είναι αυτό το πράσινο σύμφωνο που θέλετε να το φτάσετε μέχρι το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Πού θα τα βρούμε. Έχω ξανακούσει για 1,5-3 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κάνετε προβολές σε μία επταετία, αλλά όλα αυτά είναι πολύ θολά και συγκεχημένα. Επιπλέον, ε, γίνονται ακόμα διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με ανοιχτή έκβαση. Οι ήδη οι πόροι δεν είναι βιώσιμοι γιατί ε, ο φόρος στα πλαστικά εξορισμού είναι πεπερασμένος φόρος και πόρος. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ε, από την ίδια χρηματοδότηση από το αν ε, δανείζεσαι. Το ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τριπλό α, αλλά ελπίζω να μπορέσει να το διατηρήσει. Ε, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό μετάβασης, έχουμε το ταμείο αυτό που είναι ανοιχτό για όλα τα κράτη-μέλη. Από την άλλη όμως ε, υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν τραβήξει χειρόφρενο στη χρηματοδότηση. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Εγώ είμαι υπέρ της κυκλικής οικονομίας, αλλά κατά της ανακύκλωσης των υποσχέσεων και των χρημάτων. Δεν είμαστε καθόλου υπέρ της ε, δημιουργικής λογιστικής και ακόμα λιγότερο υπέρ ε, των δημοσιονομικών τυχοδιοκτικών χειρισμών. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη δράση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο ε, εξ της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς έχει ο κύριος Γιουνούς Ομαρζέ για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριοι Αντιπρόεδρε από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης η πρόοδος της Ευρώπης βασιζόταν στην εκμετάλλευση των ορυκτών μορφών ε, ενέργειας. Εκεί ε, οικοδομήθηκε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ΕΚΑΧ. Ε, είναι συνδεδεμένη με το κάρβουνο, με τον άνθρακα. Δηλαδή ο άνθρακας έχει δομήσει, διαρθρώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και σε μεγάλο βαθμό έχει συνεισφέρει στην περιφερική ανάπτυξη. Εκατομμύρια θέσεων εργασίας ήταν εξαρτημένες και σήμερα ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα καλούμαστε τώρα να κάνουμε μια πραγματική επανάσταση για να βγούμε αυτό το μοντέλο με τον όρο ακριβώς να έχουμε ως στόχο να κλείσει και το τελευταίο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο. Και λόγω της κλιματικής αλλαγής αυτό το μοντέλο έχει καταστεί απαρχαιωμένο. Όμως θα πρέπει να θέσουμε δύο προτεραιότητες πιστεύω. Πρώτον, να απορροφήσουμε το κοινωνικό κόστος και στη συνέχεια να συνοδεύσουμε τις περιφέρειες στη δίκαιη μετάβαση. Και επειδή είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ε, ε, κινητοποιηθεί πλήρως για να ανταποκριθούμε στο νομοθετικό μας έργο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόζα Νταμάτο από τους μη εγγεγραμμένους. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μία μελέτη ε, για, την, ε, για τις αλλαγές στη δική μου τη χώρα, την πόλη με στον Τάραντο. Εκεί αναφέρεται ότι δυστυχώς υπάρχει μόλυνση στην ατμόσφαιρα, στη θάλασσα και γι' αυτό η ζωή δεν είναι πλέον φυσιολογική. Έχουμε κοινωνική αποσύνθεση, ε, διαλύει το κοινωνικό ιστός. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ταμείο μπορεί να δώσει την απάντηση. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η υγεία των και δεν αρκεί ε, μία, άλλη μία μετάβαση. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε ανανέωση και ανακαίνιση των ε, εργοστασίων, όμως πρέπει να γίνουν και περιβαλλοντικές μελέτες. Η στρατηγική σημασία της Πράσινης Συμφωνίας ε, σημαίνει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να μετατραπεί σε μία πηγή έμπνευση, να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια για ανάμεσα σε ε, παράγοντε. Και τέλο, μία πρόταση. Το σύστημα τη ανταλλαγή των εκπομπών θα μπορούσε να φέρει 48 δισεκατομμύρια τα τελευταία τρία χρόνια για να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ε, χρηματοδοτηθεί και με αυτά τα χρήματα το Ταμείο τη Δίκαιη μετάβαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, εκ μέρου του ΕΛΚ, ο κύριος Νοβακόφ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί αντιπρόεδροι, ε, εγώ δεν είμαι μηχανικός αυτοκινήτων, αλλά γνωρίζω ότι η δική μας βιομηχανία είναι ίσως η καλύτερη μηχανή που υπήρξε ποτέ. Άρα δηλαδή αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να υπάρχει ένα συντονισμός για να υπάρξει ευημερία για εκατομμύρια πολιτών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν ε, προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτή τη μηχανή για σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν την βελτιώσουμε θα καταρρεύσει. Και εφόσον το γνωρίζουμε αυτό, μόνο έτσι θα πρέπει να συζητάμε για την Πράσινη Συμφωνία και για το Ταμείο της Μετάβασης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρωτοβουλία της να διασφαλίσει το μέλλον των παιδιών μας και ένα καλό περιβάλλον. Ε, βεβαίως το μέλλον δεν πρέπει να υπάρξει ζημιά στο περιβάλλον. Το μέλλον ανήκει σε πολιτικές οι οποίες δεν βλάπτουν το μέλλον των παιδιών μας. Όμως πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε πετύχουμε χωρίς να εξαφανίσουμε ολόκληρους τομείς. Μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά χωρίς να αφήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους άνεργους. Γι' αυτό λοιπόν ας εργαστούμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να απεξεργαστούμε όπως σας είπα τη μηχανή. Εγώ ανησυχώ γιατί αν έχουμε νέες καινούργιες πρωτοβουλίες θα χρειαστούμε και νέα και πολλά χρήματα και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πάρα πολύ καλή ιδέα που προβάλλεται, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις λεπτομέρειες και τις οικογένειες ε, της ε, βιομηχανίας, ολόκληρους τομείς κοινωνίας μας, να μην τους αναγκάσουμε να πληρώσουν για όλα αυτά. Ευχαριστώ λόγο στην κυρία Μπορζάν αυτή τη στιγμή, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ορίζω το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιώσιμων Επενδύσεων ως ε, σημείο κλειδί για την καινούργια Πράσινη Συμφωνία. Ε, στόχος είναι να χρηματοδοτήσει την Νέα Πράσινη Συμφωνία, αλλά να εξασφαλίσει και, άλλες, και άλλη χρηματοδότηση, να κινητοποιήσει και εθνική χρηματοδότηση, δηλαδή και χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο, δημιουργώντας ε, μια Ευρώπη πιο οικονομικά και οικολογικά πιο συνειδητοποιημένη. Ε, γνωρίζουμε την ε, προσαρμο... ότι πρέπει να προσαρμοστεί η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επίσης και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει. Ε, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουμε να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά την μετάβαση προς την ε, κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Η οδηγία για την ταξινομία είναι πάρα πολύ σημαντική και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε και του πολίτε μα. Η δίκαιη μετάβαση είναι αδύνατο να γίνει χωρίς συζήτηση με τους κοινωνικού εταίρου και με τις κοινότητες οι οποίες επηρεάζονται από τη μετάβαση. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο λόγος στην κυρία Σιλβή Μπρουινέ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένη ότι η δίκαιη μετάβαση, ε, ψηφιακή και οικολογική, μπορεί να γίνει μόνο με κοινωνική στήριξη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε απαραίτητο τους Ευρωπαίους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να περάσουν ε, σε νέους τομεί οικονομική δραστηριότητας, ε, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους. Θα πρέπει μάλιστα μεταξύ μα να μοιραστούμε τι γνώσει μα και τι εμπειρίε μα. Δεύτερον, η μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιη και σε κοινωνικό επίπεδο, να μην μείνει κανένας πίσω ή στο περιθώριο. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, την ε, ενεργειακή επισφάλεια με, ιδιαίτερη ιδιαίτερα μέτρα τιμολόγησης. Θα πρέπει η κοινωνία να δεχτεί αυτή την μετάβαση ε, προς μια κοινωνία πιο ουδέτερη κλιματικά. Πώς? Με κοινωνικό διάλογο και ε, καταπολεμώντας οποιασδήποτε ε, ε, διακρίσει, υπάρχουν και ανισότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Λάγκεν Για ένα μισή λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική περιβάλλοντος, η οικονομική πολιτική και η κοινωνική πολιτική, το να τα εξετάζει κανεί όλα από κοινό, αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ε, είναι βεβαίω απαραίτητο για να υπάρχει ε, μια δικαιοσύνη, ε, γιατί αλλιώ θα ενταθούν οι αδικίε. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο τη δίκη μετάβαση. κατ' ουσίαν η πρόταση αυτή είναι σωστή. Κυρίω οι πιο φτωχοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από την κλιματική κλιματική αλλαγή. Το δικό μας το καθήκον πρέπει να είναι να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους προστατεύσουμε κοινωνικά. Ε, Παραδείγματο χάρη, αυτό που προτείνεται για την μετεκπαίδευση των ανέργων, καλό είναι αυτό, αλλά δεν φτάνει. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την, ε, τον κοινωνικό αποκλεισμό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και εκείνου του ανθρώπου που δεν εργάζονται. Ο στόχο. Ε, της agenda της ατζέντα για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι να αντιμετωπιστεί η φτώχεια μέχρι το 2030. Να μην ενισχυθεί περαιτέρω η φτώχεια. Ο δρόμος ε, της αντιμετώπισης ε, των προβλημάτων του κλίματος πρέπει να είναι ένας, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν τα κράτη-μέλη κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων τους πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνουν και τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Και κατά τα άλλα είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε μηχανισμούς κοινωνικής υποστήριξης, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εμποδίσουμε τη φτώχεια. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να καταθέσει μια οδηγία πλαίσιο ε, για μια κατεπίγουσα πρόταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ε, σας ε, ευχαριστούμε και επόμενη κυρία Λάουρα Χιουτασάρη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι θα πρέπει να στηριχτεί η Πράσινη Συμφωνία δίδοντας κάποια κονδύλια. Αν παραμείνουμε στο επίπεδο των 100 δις, τα περισσότερα χρήματα θα διοχετευτούν στην Ανατολική Ευρώπη και αυτή η πράσινη συμφωνία θα είναι δαπανηρή για χώρες ε, όπως η Πολωνία η οποία χρησιμοποιεί κατά πολύ τον άνθρακα. Και άλλες χώρες υποδειγματικές όπως είναι η Φινλανδία θα πρέπει να περιορίσουν ακόμα περισσότερο τις εκπομπές τους. Η Φινλανδία η οποία έχει πληρώσει για τη μείωση των εκπομπών, η Φινλανδία τώρα θα κληθεί να πληρώσει για τις μειώσει σε άλλες χώρες. Στη Φινλανδία έχουμε μακρύ χειμώνα, μεγάλες αποστάσεις, η αγορά είναι περιορισμένη και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλες ε, προκλήσεις. Ε, έχουμε λοιπόν μια ε, προγραμματισμένη οικονομία η οποία επιβάλλεται σε κράτη-μέλη. Αυτή δεν έχει τίποτα να κάνει με την ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Κύριε Ραφάλσκα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλούμε για την οικολογική μετάβαση, αλλά εδώ τίθεται το θέμα της εργασίας. Ε, το κοινωνικό κόστος, το ανθρώπινο κόστος, τι θα γίνει με τους εργαζομένους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα σχέδιο που αφήνει πολύ λίγο χώρο ε, στους εργαζόμενους που απειλούνται να απολυθούν. Ιδιαίτερα εκείνοι που εργάζονται εδώ και χρόνια και είναι άνω των 50 ή των 60 ετών. Τι θα γίνει με τους εργαζομένους αυτούς που έχουν μία πείρα 30 ετών και πλέον σε συγκεκριμένους τομείς. Εδώ θίγονται η Άνω Σιλεσία, η Κάτω συλλεσία, η ε, Μεγάλη Μικρή Πολωνία, διάφορες περιφέρειες της Πολωνίας. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα κάνει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα λάβει υπόψη του αυτή την κατάσταση. Οι εργαζόμενοι αυτοί μήπως πέσουν θύματα στο βωμό της Πράσινης Συμφωνίας. Έχετε λάβει πραγματικά υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες. Εντάξει, θα τους ε, μετεκπαιδεύσετε δωρεάν, ε, θα τους κάνετε μαθήματα, φτάνει αυτό. Εδώ υπάρχουν τεράστιες απειλές. Θα αυξηθεί η ανεργία, θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα καταρρεύσουν ολόκληροι τομείς. Αυτό είναι δίκαιη μετάβαση. Αυτό θα είναι μια μετάβαση που θα δίγει τους εργαζομένους και μόνο. Κυρία Σίλβια Μόντικ από ε, την ΚΟΕ για ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι ε, ουσιαστικό στοιχείο της Πράσινης Συμφωνίας. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να μην πληγούν ε, ε, όσοι ήδη σήμερα είναι λιγότερο ευνοημένοι. Θα πρέπει βεβαίως να βοηθήσουμε τις περιφέρειες που θα θυγούν περισσότερο και όχι μόνο θα πρέπει να φροντίσουμε να μην πάνε σε λάθος τσέπες τα χρήματα αυτά. Να χρηματοδοτηθούν κυρίως οι σωστές κλιματικές ενέργειες και οι άμεσα πληγόμενοι, για να είναι ακριβώς δίκαιη η μετάβαση αυτή. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση, να μειώσουμε το κόστος και να βοηθήσουμε ε, τους εργαζομένους να μετακπαιδευτούν ε, για να αλλάξουν δουλειά, να ξεφύγουν από τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον κοινωνικό τομέα. Να συμμετέχουν όλοι στην αγορά εργασίας, γιατί αν μας ενδιαφέρει η ισότητα και η δικαιοσύνη σε όλες τις αποφάσεις μας, τότε μόνο θα έχουμε μια Ευρώπη ε, ουδέτερη προς το κλίμα, αλλά και πιο κοινωνική και μας αφορά όλους. Ο κύριος Πεντιτσίνη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να αναφερθώ και πάλι στο θέμα της Πράσινης Συμφωνίας και των Εθνικών Προϋπολογισμών. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από, τους, από την ΚΟΕ ακούσαμε ότι γίνεται λόγος για ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που θα πρέπει να χορηγείται στις κυβερνήσεις, αλλά οι κυβερνήσεις είναι εκείνες υποτίθεται οι οποίες θα πρέπει να κάνουν τις επενδύσεις. Αλλά οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν υψηλά χρέη δεν θα μπορέσουν να κάνουν επενδύσεις, πόσο μάλλον πράσινες. Αυτό λοιπόν είναι σαν παραλογισμός μακροοικονομικός, γιατί ε, οι χώρες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουν τις εκπομπές τους και κυρίως οι χώρες οι οποίες έχουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες είναι εκείνες που θα πρέπει κυρίως να κάνουν τις επενδύσεις. Εάν λοιπόν εμείς επενδύσουμε στις χώρες αυτές ε, θα μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε στην οικονομία τους ε, αλλά και στο να αντιμετωπίσουν τις εκπομπές. Οι δικές μας ε, οι εκπομπές θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη κυρίως σε σχέση με τον προπλογισμό και ας μην ξεχνάμε και τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται επόμενος ομιλητής, ε, ο κύριος Μάκους Φέπα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε εκτελεστική αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει πολύ ε, φιλόδοξους ε, στόχους για το κλίμα, οι οποίοι όμως δεν θα αυτοπραγματοθούν. Πρέπει να υπάρξουν υψηλές επενδύσεις, κάπου πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Άρα δηλαδή είναι σωστό που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει πρόταση. Αυτό το σχέδιο για τις βιώσιμε επενδύσεις δεν είναι όμως το πρώτο σχέδιο με το οποίο ασχολούμεθα εδώ στο Κοινοβούλιο. Κατά την προηγούμενη θητεία ασχοληθήκαμε με το περίφημο Ταμείο Γιούνκα και αυτό το Ταμείο μας έδωσε πολλά χρήσιμα μαθήματα για το πού πρέπει να προσέχουμε. Τρεις λέξεις κλειδί θα αναφέρω. Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει μία ισόρροπη ε, κατανομή. Ε, γιατί τα χρήματα του Ταμείου Γιούνκε τελικά ε, πήγαν εκεί που δεν έπρεπε. Δεύτερον, θα πρέπει να προσθέσουμε στο, στη σωρευτικότητα, δηλαδή δεν χρειαζόμαστε νέο προσδιορισμό ή αναπροσδιορισμό των επενδύσεων. Όχι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι επιπρόσθετες επενδύσεις. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα τελικά να έχουμε αυτή την ετικέτα, βιώσιμες επενδύσεις, αλλά τελικά να μην γίνεται τίποτα στην πράξη. Και το τρίτο που είναι σημαντικό είναι ότι πολλοί λένε οι ιδιωτικέ επενδύσει κάνουν τη διαφορά. Ναι, πράγματι, αλλά θα πρέπει να είμαστε τόσο ελκυστικοί έτσι ώστε να ε, μα στηρίξουν οι ιδιώτε επενδυτέ. Και εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε να διασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Ο στην κυρία Φρίτσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους επιτρόπους Τίμερμανς και Ντομπρόφσκης για τις προτάσεις που κατέθεσαν. Είναι όντως φιλόδοξο αυτό το σχέδιο. Είναι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που ανησυχούν βαθύτατα για το μέλλον και βλέπουν ότι έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι μια ανησυχία την οποία συμμερίζομαι. Ιδιαίτερα αν δούμε την κλιματική αλλαγή και τι σημαίνει αυτό για μας από προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μίλησε για μια κοινωνικά ισχυρή Ευρώπη και έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες αγωνιζόμαστε ανέκαθεν πάρα πολύ για τον κοινωνικό πυλώνα. Το 2017 έγινε αυτό πραγματικότητα στη Σουηδία, στο Γκέτεμπορκ. Και αυτός ο κοινωνικός πυλώνας θα είναι αποφασιστικότατος για τη νέα Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους, χρειαζόμαστε καλές θέσεις εργασίας για άνδρες και γυναίκες με καλή εκπαίδευση, με καλές δεξιότητες και προσόντα. Παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μισθούς και ημερομίσθια για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν από αυτούς. Εγώ που είμαι Σουηδή θα προτιμούσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να κυριαρχήσει το βορειοευρωπαϊκό μοντέλο, το σκανδιναβικό μοντέλο. Θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες φυσικά ε, πολύ στενά. Και αυτό που έχει σημασία είναι να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών στην Ευρώπη. Ας αρχίσουμε από κοινού αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Καταλίν Τσέχ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι ότι θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό του τους πολίτες, όχι σε κυβερνήσεις ούτε τις εταιρείε. Η δίκαιη μετάβαση θα πρέπει να φτάσει μέχρι τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης. γιατί εκεί η βοήθεια μπορεί να αποτελέσει διαφορά ανάμεσα στο πεθαίνω στο κρύο ή με ζεστό στο χειμώνα. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Δεν θα πρέπει να επωφεληθούν από τις ε, κοινοτικές αυτές ενισχύσεις προκειμένου να πλουτίσουν τους φίλους τους. Θα πρέπει η βοήθεια αυτή να δοθεί με διαφάνεια και με σωστά εργαλεία διαχείρισης. Διαφάνεια και αλληλεγγύη θα πρέπει να χαρακτηρίσουν την όλη διαδικασία η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα δεν θα είναι εύκολη, ε, αλλά χωρίς αυτά δεν μπορεί να πετύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο λόγος στον κύριο Άικχαουτ για ένα μισή λεπτό. Όταν παρουσιάσατε την Πράσινη Συμφωνία το Δεκέμβριο, ήταν σαφέ ότι πρόκειται για μια αλλαγή, για μια καινούρια κομισιόν, με καινούρια εστίαση, καινούριε προτεραιότητε. Το στηρίξαμε πλήρω και το στηρίζουμε ακόμα. Όμω το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι, θα γίνουν πραγματικά επενδύσει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για μια ελάσσονο σημασία αλλαγή, πρόκειται για μια μετάβαση σε όλε τι περιφέρειε, σε όλε τι χώρε, σε όλου του κλάδου οικονομία. Και αυτό απαιτεί επενδύσει. Και εκεί Πρέπει να πω, δεν μπορώ να βγάλω οριστικό συμπέρασμα γιατί δεν έχω δει την τελική πρόταση, αλλά από τις πρώτες εκδοχές που βλέπω είναι ότι έχουμε ε, καινούρια πράσινη συμφωνία ε, χωρίς να έχουμε απαραίτητα καινούριο πλαίσιο για επενδύσεις. Σαν να κάνουμε την ίδια συζήτηση που κάναμε και από την προηγούμενη Κομισιόν για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Όταν μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιώσιμων Επενδύσεων, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δεν θα είναι ένα ακόμα ε, ε, πρόγραμμα, σχέδιο Juncker 2,1, 2,2, 2,3. Θα πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη θεμελιώδη αλλαγή. Είναι δυνατόν. Αν δούμε τι πράσινε κρατικέ προμήθειε, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή, να κάνουμε τη διαφορά. Και θα πρέπει όμω να αλλάξουμε και τη φορολογική μα πολιτική τις φορολογικές μας πολιτικές. Κάτι λέτε για αυτό το θέμα, αλλά είναι τόσο πολύ έμεσο αυτό που λέτε ότι ίσως στο τέλος αυτού του διαλόγου να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που κλπ. κλπ. Δεν μας πείθει αυτό. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Νταβίτ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα όλου του πλανήτη εμείς εδώ από μόνοι μας. Είναι αδύνατο αυτό. Κυρία Φόντερ Λάγεν, είναι γιατρός από όσο ξέρω. Όμως, ε, η βασική αρχή για τους γιατρούς είναι να μην βλάπτουν τους ασθενείς τους. Ε, κατά την άποψή μου η Πράσινη Συμφωνία δεν είναι καλά προετοιμασμένη, ούτε είναι δυνατόν να εφαρμοστεί έτσι όπως έχει. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να πάρουμε τα λεφτά από τους πλούσιους και να ε, θεραπεύσουμε αυτόν τον τρόπο τους φτωχούς. Ε, είδαμε τι έγινε με τέτοιου είδους φιλόδοξα σχέδια στο παρελθόν όταν δεν είχαμε εξετάσει επαρκώς τις συνέπειε και φοβάμαι ότι ε, τα σχέδιά σα αυτή τη στιγμή είναι θολά και βασίζονται απλώς σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση. Το Σενόφσκι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Εποσχέσεις ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενεργειακή πολιτική, πολύ φιλόδοξη η στόχη και πολύ σαφής. Ο δρόμος όμως προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον θα πρέπει να σημάνει ότι δεν θα μείνουν πίσω οποιασδήποτε περιφέρειες σήμερα εξαρτώνται από τον άνθρακα. Χαίρομαι που κάνει την πρόταση για το συγκεκριμένο ταμείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να μετασχηματιστεί και η οικονομία ε, συνήθως είμαι επιφυλακτικός όταν βλέπω τους υπολογισμούς που γίνονται επί χάρτου. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται όντως επενδύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, δισεκατομμυρίων επενδύσεις σε όλη την Ένωση. Χρειάζεται μια σωστή μελέτη αντικτύπου για να ξέρουμε τι θα σημάνει αυτό για κάθε περιφέρεια. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνδέομαστε πολύ με το Ταμείο Συνοχής φοβάμαι ότι θα υπάρξουν μεγάλες εντάσεις εκεί, όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και μεταξύ περιφερειών. Ευχαριστώ. Νικολάη Βίλουμσεν. Ένα λεπτό παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε πρόσφατα ε, να αποδυναμώνει μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να αποδυναμώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συλλογικέ συμβάσεις. Χαίρομαι που ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να αναγνωρίζει ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις αυξανόμενες ανισότητες. Γίνεται μια πρόταση τώρα για ένα κατώτατο ε, ημερομίσθιο αυτή είναι πολύ λάθος πρόταση. Φοβάμαι ότι θα είναι άλλο ένα ράπισμα προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων. Ας φτιάξουμε ένα κοινωνικό πρωτόκολλο που να βάζει πάνω από την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. και να σταματήσουν οι διάφορες λαμογές στις δημόσιες προμήθειες ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση για να σταματήσει η ομή εκμετάλλευση των ξένων εργαζομένων και των ξένων συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ρόουλαντ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα κρίσιμο σημείο όπου βλέπουμε να καταστρέφονται θέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της Πράσινης Συμφωνίας. Αυτή η υπόσχεση περί δίθεν θέσεων απασχόλησης, αυτό ήταν μια αυταπάτη ε, και υπήρχε λάθος άποψη ότι υποτίθεται θα προέκυπτε ευημερία. Αλλά αυτοί όλοι οι γραφειοκράτες ποτέ δεν συνέστησαν, δεν σύστησαν μια επιχείρηση, δεν ξέρουν ποια είναι η βιομηχανική βάση στην Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για μια καταστροφή. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ήδη ότι θα χαθούν 40.000 ε, θέσει απασχόλησης λόγω των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και αυτά που λέτε εδώ για την στην συμφωνία μου θυμίζουν από αυτά που έλεγαν Αμερικανοί, ότι για να σωθεί ένα χωριό πρέπει πρώτα να το καταστρέψει. Ε, το ίδιο, την ίδια λογική έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποτίθεται έχει τη δύναμη να φτιάξει θέσει απασχόληση, αλλά πρώτα θα καταστρέψει αυτέ που υπάρχουν. Τα 30 δι ευρώ υποτίθεται θα βοηθήσουν Πολωνία, Τσεχία. Εγώ προβλέπω ότι ο αριθμό θα τριπλασιαστεί γιατί η Κομισιόν ε, θα πληρώσει γι' αυτό το την τρελή πράσινη συμφωνία ε, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή την απαρχιωμένη βιομηχανική βάση σκόπιμα την κατέστρεψαν. Έχουμε μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε παρακαλώ. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Αν ε, δεν την δέχεστε παρακαλώ επόμενος ομιλητή, ε, ο κύριο ε, Νίκο Τινίνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ πολύ καλά ότι δεν είσαστε και απόλυτα ικανοποιημένοι, ε, διότι η κυβέρνηση σα αφήνει τους ανθρώπους εγκατρελειμμένου. αλλά ε, κατ' ουσίαν γιατί έρχεστε εδώ. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μένετε στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί ήσασταν και εκεί να παραμείνετε. Την απάντηση παρακαλώ στη μπλε κάρτα. Σα ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό ήταν ερώτηση, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να σας απαντήσω. Παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το κοστο ήταν ένα ένα-τρει. λίρε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εμείς κάναμε αυτή, αυτόν τον υπολογισμό και εδώ πριν ε, υπογράψετε θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Τίμερμανς ε, τι θα σημαίνει το κόστος από το να χαθούν όλες αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Τώρα εμείς 12 εκατομμύρια λίρες το χρόνο πληρώνουμε για τι διάφορες πράσινες εισφορές. Ε, είναι λοιπόν ένας φόρος τον οποίο καλούνταν να το πληρώσουν οι πιο φτωχοί. Πολύ ωραία. Επόμενος ομιλητή, ο κύριος Ντένι Ράτκε για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Αντιπρόεδρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και για την αρχή που κάνατε σήμερα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν περιμένουμε τίποτα άλλο παραπάνω. Και τα λέω αυτά, έχοντας κατά νου τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να ξεφύγουμε λιγάκι από τα συνθήματα. Να ξεφύγουμε από αυτό το θολό τοπίο, γιατί έχει τελειώσει η προεκλογική εκστρατεία και για εσάς, κύριε Τίμερμανς. Άρα, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό πλέον να μην παραμένουμε στο κατά προσέγγιση, αλλά πολύ συγκεκριμένα να λέμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει και για το θέμα της κοινωνικής Ευρώπης. Το θέμα του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβαση το χαιρετίζω ανεπιφύλακτα, αλλά αυτό που δεν πρέπει να συμβεί είναι συνθήματα του προϋπολογισμού ε, και κονδύλια ακόμα να μεταφέρονται, απλά να πηγαίνουν στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, γιατί στην περίπτωση αυτή οι άνθρωποι που δουλεύουν στη βιομηχανία, οι άνθρωποι αυτοί λόγω των αλλαγών ε, και της κλιματικής αλλαγής κινδυνεύουν. Και αυτούς να τους βάλουμε να τσακώνονται με μακροχρόνια άνεργους που έχουν άλλα προβλήματα. Να μην βάλουμε τους αδύναμους της κοινωνίας να τσακώνονται μεταξύ τους. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί πρέπει να πούμε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να οδηγήσει σε ε, καταστροφή δομών. Και για να το πετύχουμε αυτό να δημιουργήσουμε νέο πλούτο, όχι να μεταφέρουμε τα χρήματα από τη δεξιά στην αριστερή τσέπη. Η κυρία ε, εξακολουθεί να υπάρχει σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά ε, το κατά πόσον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητε και την κλιματική αλλαγή μαζί. Και το Ταμείο Δίκαιης ε, Μετάβασης ε, γι' αυτό υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο προβλήματα μαζί. Υπό την βέβαια ότι υπάρχει αποφασιστικότητα και βούληση. Η νέα πράσινη συμφωνία θέλει να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρο προς την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας, ταυτόχρονα όμως χωρίς να αφήσει πίσω ή εκτός τους πιο ευάλωτους. Αναγνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα του άνθρακα χρειάζεται να προστατευτούν προκειμένου να, αποφελ, να από αυτή τη μετάβαση. Γιατί τελικά οι αυριανέ θέσει εργασία θα χρειαστούν άλλου τύπου δεξιότητε και θα πρέπει το εργατικό μα δυναμικό να προσαρμοστεί ενώ προετοιμάζονται και καινούριε γενιέ. Ε, οι πράσινες πρακτικές, ε, οι υπηρεσίες και αγαθά δεν θα πρέπει επίσης να ε, αποκλείουν ένα κομμάτι του πληθυσμού. Θα πρέπει η κοινωνία να συμμετάσχει και οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, που επηρεάζονται, οι κοινότητε ε, που επηρεάζονται θα πρέπει να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό, θα πρέπει να στηριχτούν, να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι και να δημιουργηθούν καινούριε θέσει εργασία οικολογικέ, πράσινε ε, και βιώσιμε με ανανέωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Χρειάζεται βέβαια απαραίτητη χρηματοδότηση και απαραίτητε πολιτικέ. Με αυτέ τι προποθέσει μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούριε θέσει εργασία σε μια καινούργια οικονομική πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει Πρόεδρο, συγγνώμη. Δίνω το λόγο στην κυρία Αρμό. Κύριε Πρόεδρε, ε, οι κοινωνίες ε, της Ανατολικής Ευρώπης ε, είναι σε θέση για να μιλήσουν για την οικολογία γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη σχέση και δεσμούς με το περιβάλλον και με τη γη τους. Οι αλυσίδες παραγωγής είναι πολύ πιο κοντά στην κοινωνία επίσης. Έχουμε πολλά παραδείγματα μετάβασης ήδη σε περιοχές που εξαρτώνται κατά πολύ από τον άνθρακα στο παρελθόν και που τώρα επωφελούνται ε, και χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει οι πολιτικέ μα να είναι σαφείς, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο τρόπο. Χρηματοδότηση, συνδρομή για την υλοποίηση σχεδίων, η αναγνώριση διαφόρων ενεργειακών μειγμάτων, ε, προσαρμοσμένων στην κάθε χώρα, προκειμένου να μην δώσουμε τροφή στους ευρωσκεπτικιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Νίνιστρο. Για ένα λεπτό. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. There you go. Madam President, the Green Deal is the most ambitious... Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το πιο φιλόδοξο σχέδιο τις τελευταίες δεκαετίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να δούμε ότι επηρεάζει όχι μόνο του Ευρωπαίου πολίτε, αλλά και τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Είναι μια ευκαιρία προκειμένου να βρεθούμε σε μια ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουμε έναν θετικό οικονομικό κύκλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταφέρουμε επίση να εξάγουμε τεχνογνωσία. Το θέμα είναι ότι η πρόταση που έχουμε ενώπιό μα αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ασαφή. 5 δισεκατομμύρια μόνο βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι δεσμεύονται. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ασαφεί προτάσει. Και πέρα από το ποσό αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι περαιτέρω δράσει θα πρέπει να αναλυφθούν ούτω ή άλλω. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ας μην ξεχνάμε ότι ε, και αυτή με τη σειρά της μπορεί να μοχλεύσει περισσότερες επενδύσεις και μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να έρθουν να προσθεθούν και ιδιωτικά κεφάλαια στα δημόσια κεφάλαια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένες πλέον ε, προϋποθέσεις προκειμένου να μπορούμε να προωθήσουμε πραγματικά μια πράσινη οικονομία απομακρυνόμενη όλο και περισσότερο από τα ρηκτά καύσιμα. Σε εύχομαι καλή τύχη βέβαια στο χείρημά σας αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Ραήλ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, συζητάμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία σαφώς θα επηρεάσει πάρα πολύ τις περιοχές οι οποίε εξαρτώνται από την εξόριξη άνθρακα. Τα τελευταία 33 χρόνια ασχολήθηκα με όλες αυτέ τι περιοχέ που παράγουν άνθρακα. Στις περιοχές βέβαια αυτές πλέον δεν βλέπουμε να υπάρχουν ούτε πολλοί πολίτε ούτε σημαντικά δείγματα οικονομίας. Ακόμα και από την ε, περιοχή της Γερμανίας που κάταγω εγώ έχουμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό πλέον απασχόλησης. Στις ε, περιοχές επίσης που παρήγαν άνθρακα στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στο Μένο Βασίλειο η κατάσταση είναι παρόμοια. Και το ίδιο ακριβώ βλέπουμε και στην Πολωνία, όπου θα χαθούν σίγουρα εκατοντάδε χιλιάδε θέσει απασχόληση. Μιλάμε λοιπόν για μια επερχόμενη καταστροφή που δεν έχει να κάνει μόνο με τι περιοχέ εξόριξη άνθρακα, αλλά και με τι περιοχέ τη αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουμε συμβούλου στα πλαίσια τη γερμανική κυβέρνηση που μα λένε ότι και στον τομέα αυτό θα χαθούν επίση πάρα πολλέ θέσει απασχόληση. Α σταματήσουμε λοιπόν την απόλυτη αυτή τρέλα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Ξέγκο Τομπισόφσκι για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μέρημνα για το κλίμα είναι πολύ σημαντικό και υπεύθυνο έργο. Για να δημιουργήσουμε μια πράσινη, μια οικολογική τάξη, θα πρέπει να δούμε ε, σε ποια θεμέλια θα στηρίζεται αυτή η πράσινη τάξη. Γι' αυτό έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη, πρόκειται να έχει διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη για το πόσα χρήματα θα, χρειαστούν τι κονδύλια για επενδύσεις ώστε να πραγματοποιήσουν αυτή την ενεργειακή μετάβαση αποτελεσματικά και για να μην δημιουργηθεί ενεργειακό χάσμα στην Ευρώπη. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο χρόνος θα χρειαστεί αυτό το πρασίνισμα των οικονομιών των μεμονωμένων χωρών. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, υπολογίζουμε ότι το συμπληρωματικό κόστος αυτής της αλλαγής θα ανέλθει στο 2,6 ως 4,3 του ΑΕΠ για τα έτη 2020-2050, δηλαδή πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι επιβάρηση 1,7 έως 2,3 φορές περισσότερη από την επιβάρηση του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στην Πολωνία έχουμε την Σιλισία που έχει ανθρακοριχεία και εξαρτάται από τον άνθρακα. Ε, υπολογίζεται ότι στον τομέα του άνθρακα απασχολούνται περίπου 200.000 εργαζόμενοι και το μέσο κόστος αντικατάστασης ενός ε, μιας θέσης εργασίας είναι περίπου 250.000 ευρώ. Πώς λοιπόν θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη νέα πράσινη τάξη, θα πρέπει όλοι να έχουμε ισότιμες ευκαιρίες. Στα, στα πλαίσια της ε, γαλάζιας κάρτας κάποιος συνάδελφος θέλει να σας υποβάλει ερώτηση. Ο κύριος Πέτρας ο κύριος Πέτρος Κόκαλης έχει μια ερώτηση να σας υποβάλει. Παρακαλώ. Ο συνάδελφος γνωρίζει τι επίπτωση ε, θα έχουν στο ΕΠ ποσοστιαία οι κλιματικές αλλαγές και η υπερθέρμανση του πλανήτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τομπισόφσκι για μισό λεπτό για την απάντησή του. Αυτό δεν το αφισβήτησα στην δική μου παρέμβαση. Απλώς και μάλιστα είπα ότι η μέρημνα για το κλίμα αποτελεί τεράστιο και υπεύθυνο έργο. Για να ανταπεξέλθουμε όμω σε αυτό το έργο θα πρέπει να έχουν προηγηθεί διεξοδικέ αναλύσεις ώστε να λάβουμε υπόψη την προστασία του κλίματος, αλλά ταυτόχρονα την προστασία του ανθρώπου και των θέσεων απασχόληση. Δεν είμαι κατά του προγράμματο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προσβλέπει να γίνει παγκόσμιο ηγέτη σε θέματα περιβαλλοντικά, θα πρέπει να έχει κάνει του απαραίτητου προπολογισμού για να διαφυλάξουμε και τι πρώτε εργασίε. Ο κύριος Γκουσμάου, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε με τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης θα πρέπει να είναι δίκαιο και η Νέα Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να είναι κοινωνική. Αυτό όμως δεν θα καταστεί δυνατό αν οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι έρχονται σε ανταγωνισμό με άλλες πολιτικές και περικόπτονται τα κονδύλια τους. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μην ε, μεταφέρουμε κονδύλια από το ένα τμήμα στο άλλο τμήμα του προπολογισμού. Ε, ε, και νέα κονδύλια να προβλέπουμε μόνο για την στρατιωτικο ε, μιλιταριστική μας ιδεολειψία και όχι για τις παλιές πολιτικές. Ε, είπατε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι όμως χρήματα που θα ε, επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε ξέρει αν θα προσελκύσει αυτά τα κονδύλια από άλλου για να επενδυθούν. Ούτε γνωρίζουμε αν θα είναι πραγματικά κοινωνική η νέα πράσινη συμφωνία. Γιατί αν ε, στερήσουμε από τις περιφέρειες συνοχής τα κονδύλια, από περιφέρειες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κλιματικών αλλαγών τα κονδύλια, τότε δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τη νέα δίκαιη μετάβαση. Ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο με αυτό το επενδυτικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα και το Ταμείο Δικής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγαμε ανέκαθεν ότι οι νέε προτεραιότητε θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από συμπληρωματικού πόρου, επιπρόσθετου. Και είναι πολύ θετικό που το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση έχει 7,5 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ πρικοδότηση. Η ερώτησή μου είναι, αρκούν αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δίκαιη μετάβαση. Αυτό θα πρέπει να μελετήσει και να εξακριβώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον και η συμπληρωματικότητα είναι κάτι θετικό. Συμπληρωματικότητα με την πολιτική συνοχή. Θα πρέπει όμω οπωσδήποτε η πολιτική συνοχή να μην αλλοιωθεί. Η δίκαιη μετάβαση σε καμία περίπτωση δεν θα λάβει χώρα ε, εις βάρος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Επιπλέον θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να προσδιορίσουν τα επενδυτικά του σχέδια. Θα πρέπει να ξέρουν τι θέλουν για τις περιφέρειές τους. Είδε μη, τα κονδύλια που έχουν προσδιοριστεί ε, για κάθε περιφέρεια θα μείνουν αχρησιμοποιητά και θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες και θα, θα μας λένε στις Βρυξέλλες ότι το τα κράτη-μέλη δεν ήξεραν τι ήθελα. Θα πρέπει κάθε περιφέρεια και κάθε χώρα μέλος να κάνει τη δουλειά του, να αναλάβει τις ευθύνες του στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιμώνα Μποναφέ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χίλια δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή μας λέτε για τα επόμενα δέκα χρόνια ως βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό είναι ο σημαντικότατος στόχος που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου το 2050 να γίνουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με κλιματικά ουδέτερη και χωρίς αποκλεισμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερους σπόρους σίγουρα. Αν πραγματικά όμως θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, θα χρειαστούμε ακόμα περισσότερους σπόρους ως προς την πρόταση όμως Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο καινοτομίες βλέπω αυτή τη στιγμή. Πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το Ταμείο δίκαιη μετάβαση, το οποίο να επιτρέψει όντω ορισμένε περιφέρειε οι οποίε βασίζονται ακόμα στο ρηκτά καύσιμα να καταφέρουν να περάσουν στην ε, νέα, στο νέο αυτοκλιματικό οικολογικό καθεστώς. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεύτερον, όσον αφορά το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη. Θα πρέπει εδώ πέρα οι επενδύσει που θα γίνουν να μην συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του δημοσίου ελλείμματο